δικές εκλογές για να μπορούν οι πολίτες της Βενεζουέλας να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση. Ευχαριστώ, Ίντσερ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ως σοσιαλδημοκράτης είμαι πεπισμένη ότι οι πραγματικά ισότιμες κοινωνίες όπου υπάρχει ειρήνη και ελευθερία ε, πρέπει να παρέχουν πρόσβαση και στα δημοκρατικά δικαιώματα και στις κοινωνικές ελευθερίες. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή Κοιτώντα κανεί τη Βενεζουέλα, βλέπουμε ότι οι πολίτε φεύγουν από τη χώρα γιατί ε, δεν έχουν ε, τίποτα τα παραπάνω. Πάνω από 4,5 εκατομμύρια Βενεζολάνοι πολίτε έχουν φύγει από τη χώρα. Όλο ένα και περισσότεροι φεύγουν κάθε μέρα. Η υπάτη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες έχει ανακηρύξει αυτή την κατάσταση ως μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές καταστροφές στον κόσμο. Θα πρέπει πλέον οι πολίτες της Βενεζουέλας να ε, ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Πρέπει να απαιτήσουμε την διεξαγωγή δίκαιων και ελεύθερων εκλογών, θεμελιώδη δικαιώματα, πρόσβαση στις θεμελιώδεις ελευθερίες ε, για όλους και να αυξήσουμε και την ανθρωπιστική μας βοήθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Μπιλμπά Μπαραντίκα. Πίνια, λοιπόν. Ευχαριστώ. Η Διεθνής Διάσκεψη Ελεγγύης της Βρυξέλλας ε, έλαβε ε, αριθμού σε σχέση με το κόστο που έχει η δικτατορία του Μαδούρου στου Βενεζολάνου. Ε, πάνω από 4,5 εκατομμύρια άνθρωπα ήδη έφυγαν από τη, μιζέρια, από τη μιζέρια και την ανασφάλεια. Το 2020 μπορεί να φτάσουν τα 6 εκατομμύρια. Το 80% φεύγουν σε γειτονικέ ε, χώρες. Όμως παρόλα αυτά έχουμε ξενοφοβικού λόγου και υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη πίεση σε μια κρίση η οποία αντιμετωπίζεται με περισσότερο με δεσμεύσει παρά με κονδύλια. Γι' αυτό είναι επίγον να με τα κονδύλια που πρέπει να δοθούν στα θύματα και να τηρήσει κανείς ε, τις ε, δεσμεύσεις του. Ε, όμως ε, χρειάζονται πιο συγκεκριμένες λύσεις που θα επικεντρώνονται στο να βοηθηθούν οι Βενεζολάνοι στη χώρα τους. Θα πρέπει να τεθεί τέλος στο πολιτική εμπλοκή που προτείνει ένα καθεστώς που θα δημιουργήσει, θα οδηγήσει σε ελεύθερες εκλογές και πρέπει να υποστηριχθεί αυτό από την Ένωση. Σας ευχαριστώ, κύριε Κέμπα, για ένα λεπτό. Κύριε Κέμπα. Δεν είναι εδώ. Ο κύριος Ντέβιντ Λέγκα, για ένα λεπτό. Ο κύριος Ντάβιτ Λέγκα, για ένα λεπτό παρακαλώ. right. Thank you, Chair. Ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Μπορέλ. Σε ό,τι αφορά την κρίση στη Βενεζουέλα και την συζήτηση που κάναμε τον Ιούλιο, επενθύμησε το Κοινοβούλιο ότι οι Βενεζολάνοι πεθαίνουν από την πείνα σε μια χώρα που στο παρελθόν ήταν τόσο πλούσια. Παραμένει λοιπόν αυτό το γεγονό. Και μάλιστα οι Βενεζολάνοι πυροβολούνται από τι ε, αρχέ ε, του Προέδρου Μαδούρο. Και οι πολίτες που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη χώρα περνούν από πολύ δύσκολα μονοπάτια, δεν έχουν τα απαραίτητα έγγραφα και έτσι δεν έχουν και πρόσβαση σε θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό τους καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους ε, σε, στους διακινητές, στους ε, στα διάφορα κυκλώματα πορνεία και διακίνηση ανθρώπων και το καθεξής. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερε προσφυγικέ ε, κρίσεις τη της εποχής μας. Ε, γι' αυτό και ζητώ την ε, ε υλοποίηση όλων των υποστηρικτικών μέτρων της Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόμα και με το πάγωμα περισσοκών στοιχείων. Και όσοι εδώ στο Κοινοβούλιο συνεχίζουν να στηρίζουν το Μαδούρο και αντιτίθενται στι ε, ενέργειέ μα να βοηθήσουμε του Βενεζολάνου, είμαι σίγουρη ότι θα έχουν την θέση που του αξίζει στην κόλαση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ανδρουλάκης, για ένα λεπτό. Πάνω από 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τη Βενεζουέλα λόγω της απελπιστικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία της ύπατης αρμοστίας του οηε για τους πρόσφυγες ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί ραγδαία στα 6,5 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2020. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες μετακινήσεις πληθυσμού στην εποχή μας. Η κατάσταση αυτή δεν επιτρέπει την επιβολή γενικών οικονομικών κυρώσεων γιατί μπορεί να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο η ανθρωπιστική κρίση. Οι όποιε κυρώσει πρέπει να είναι στοχευμένε σε πρόσωπα που φέρουν την ευθύνη για τη σημερινή τραγωδία το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο οφείλει να προκρίνει μια πολιτική λύση που θα οδηγήσει σε ελεύθερες δημοκρατικές εκλογές με την παρουσία διεθνών παρατηρητών ως το πρώτο βήμα της ομαλοποίησης. ο αυταρχισμός τα βασανιστήρια και η εξοθλίωση ενός λαού με όποιο περιτύλιγμα και αν παρουσιάζονται στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο είναι αδιανόητο να βρίσκουν υποστηρικτές ανάμεσά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Μια γαλάζια κάρτα. Ο κύριος Σόκολ θα ήθελε να σας υποβάλει ένα ερώτημα. Το δέχεστε? Δέχεστε την ερώτηση? Μπορείτε να βάλετε τα ακουστικά σας. Κύριε Ανδρουλάκη. Κύριε Ανδρουλάκη, Δέχεστε μπλε κάρτα από τον κύριο Σόκολ. Ωραία. Κύριε Σόκολ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που επιτέλους άκουσα κάποιον από τη αριστερή πλευρά του Κοινοβουλίου να μιλήσει κάτι για τις ε, αιτίες ε, των όσων συνέβησαν. Το ερώτημα μου είναι, τα καθεστώτα του Τσάβε και του Μαδούρο είναι αυτά που είναι υπεύθυνα για την πείνα και την κρίση στη Βενεζουέλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο, κύριε Ανδρουλάκη, για να απαντήσετε. Για 30 δευτερόλεπτα. Η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα και σε άλλες χώρες μας κάνει να καταδικάζουμε τέτοια φαινόμενα όποιοι και αν είναι υπεύθυνοι. Εμείς δεν βάζουμε σε ζυγαριά ούτε χρωματίζουμε τον πόνο των ανθρώπων και όλες αυτές τις τραγωδίες. θέλω να υπογραμμίσω ότι είναι προφανές ότι οι ευθύνες του κύριου μαδούρο είναι αυτές που οδήγησαν σήμερα να είναι σε μια τραγική κατάσταση ο λαός της βενεζουέλας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ζόφκο για ένα λεπτό. Um, Αξιότιμα μέλη. Κύριε Πέτα πριν από δύο λεπτά δώσαμε το βραβείο Σαχάροφ στην δημοκρατική αντίσταση τη Βενεζουέλα και αποστήλαμε πολύ ισχυρή προειδοποίηση προ του ηγέτε αυτή τη χώρα να αλλάξουν προκειμένου να εκδημοκραστεί πραγματικά η χώρα. Δυστυχώ ε, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και γινόμαστε μάρτυρε μια ανθρωπιστική ε, κρίση. 4,5 εκατομμύρια Βενεζολάνοι έχουν φύγει από τη χώρα το 2015. Και αν συνεχιστεί αυτή η τάση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα φτάσουμε στα 6,5 εκατομμύρια ενδεχομένως μέχρι το 2020. Η κατάσταση δεν μπορεί να επιληθεί χωρίς ε, την παρέμβαση της ευρύτερης διεθνούς κοινότητα. Γι' αυτό και υποστηρίζω τις ε, προσπάθειες της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Κομισιόν για να έχουμε ε, ελεύθερες και δίκαιες εκλογές και σωστή κατανομή των εξουσιών. Θα πρέπει να αποκατασταθεί η δημοκρατία και θα πρέπει να υπάρχει αυτό το, το σύστημα του δημοκρατικού ελέγχου. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τζούλι Βόρντ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Η προσφυγική κρίση της Βενεζουέλας ε, θεωρείται ότι είναι η χειρότερη προσφυγική κρίση το 2020 και είναι αυτή που δέχεται τη μικρότερη χρηματοδότηση στην ιστορία και δεν φιγουράρει καν στις, ε, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Βενεζουέλα είναι δεύτερη μετά τη Συρία σε σχέση με τον αριθμό των εκτελεσμένων ανθρώπων που ζουν εκτός ε, της πατρίδας τους. Όμως, η Πατερμοστία προβλέπει ότι περίπου 6,5 εκατομμύρια Βενεζουλάνοι θα ζουν εκτός της χώρας τους μέχρι το 2020 και αν θα ξεπεράσει ε, τον αριθμό των εκτοπισμένων ε, στη Συρία. Αυτή η κρίση πλήττει εκατομμύρια πολίτες ε, και έχουμε 17 χώρες υποδοχής. Συνήθως είναι ηλικιωμένοι οι γυναίκες και τα παιδιά οι οποίοι στερούνται τα περισσότερα, συχνά είναι πεινασμένοι και άρρωστοι και επίσης οι γυναίκες γυναίκες ε, κινδυλεύουν από την πορνεία, το είναι σωματική βία και την εμπορία ανθρώπων και τη σεξουαλική κακοποίηση. Φοβούνται ε, φυσικά και δεν αναφέρουν αυτά τα περιστατικά. Οι γυναίκες, ε, οι νέοι και οι μειονότητες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην εξέβρεση βιώσιμων λύσεων για την ειρήνη και τη σταθερότητα και εμείς ως Ευρωπαίοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε έκκληση για στρατιωτική παρέμβαση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σόκολ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία ε, Πρόεδρε. Είναι απίστευτο. Ακούμε δικαιολογίες και ακούμε και κάποια σχετικοποίηση του ποιος φέρει πραγματικά την ευθύνη. Έχουμε ένα ε, εγκληματικό κομμουνιστικό καθεστώς, ε, πρώτα του Τσάβες ε, και μετά του Μαδούρο. Ο Τσόρτσιλ είχε πει ότι οι σοσιαλιστές ε, παράγουν φτώχεια, ισόνομα και ισότιμα κατανεμημένοι. Βλέπουμε τώρα ότι στην Βενεζουέλα ελέγχονται τα πάντα, ελέγχονται οι τιμές και το αποτέλεσμα είναι ότι την τελευταία δεκαετία στη Βενεζουέλα η παραγωγή τροφίμων έχει μειωθεί κατά 75% γιατί το κράτος ελέγχει τα πάντα. Χρησιμοποιούνται σοσιαλιστικές μέθοδοι που έχουν αποδειχθεί ότι είναι αναποτελεσματικές. Εκατομμύρια ανθρώπων εγκαταλείπουν τη Βενεζουέλα και στο μέλλον έχουμε ακόμα περισσότερους. Έχουμε το έγκλημα, έχουμε τους υπέτειους, είναι το κομμουνιστικό καθεστώς. Ας μην επιτρέψουμε να επαναληφθούν τέτοιου είδους καταστάσεις. Για ένα λεπτό, ο κύριος Λιμπεράτσκι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία, κύριε είπατε εκπρόσωπε, είναι δύσκολο, ήταν πριν από κάποια χρόνια δύσκολο όταν ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια της Βενεζουέλας ήταν δύσκολο να προβλέψει κανείς ε, το τι θα ακολουθούσε, ε, το τι θα προσέφερε ο λαϊκισμός για να επιβιώσει. Και τώρα έχουμε κακή διακυβέρνηση αφενός και φτώχεια και ε, πόνο των πολιτών από την άλλη. Και μπροστά μας έχουμε και ένα δίλημα να επιβάλλουμε κυρώσεις εγώ συμφωνώ μαζί σας κύριε είπατε εκπρόσωπε ή μήπως θα πρέπει να προτείνουμε κάποια λύση παραδείγματο χάνει πετρέλαιο, σαντάλλαγμα χρημάτων, ε, ενδυμάτων. Εγώ θα έλεγα ναι βεβαίω, ναι γιατί όχι γιατί έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και αυτό είναι το σημαντικότερο. Ευχαριστώ. Κύριε Σάντο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα ε, πήρε δραματικές διαστάσεις. Είναι χαρακτηριστικά τα νούμερα. Το 90% του πληθυσμού ζει κάτω από το κατόφλι της φτώχειας. Πάνω από το 50% των παιδιών δεν πάνε στο σχολείο. Μέχρι σήμερα ε, έχουμε πάνω από 4,5 εκατομμύρια εκτοπισμένους και προβλέπεται ότι ε, αυτό το αριθμό, αν δεν επιληθεί η κρίση, μπορεί να φτάσει και τα 10 εκατομμύρια εκτοπισμένους μέχρι το 2023. Φανταστείτε ότι αυτός ο πληθυσμός μπορεί να συγκριθεί με όλο τον πληθυσμό της Πορτογαλίας. Το Διεθνές Οικονομικό Πρόγραμμα Υποστήριξης των Προσφύγων ε, δεν υλοποιείται. Έχει καθυστερήσει και φαίνεται ένα αποτελεσματικό μπροστά στην σοβαρότητα της κατάστασης και στις ε, αναγκαιότητες των εκτοπισμένων, στις ανάγκες των εκτοπισμένων. Όμως ε, δεν θα αρκέσει όποια οικονομική στήριξη και να δοθεί. Χρειάζεται να βρούμε μια οριστική λύση που να επιτρέπει να υπάρξει σταθερότητα στη χώρα. Και αυτό θα είναι δυνατό αν αναγκάσουμε τους ε, πολιτικούς να βάλουν το συμφέρον της χώρας πάνω από το ατομικό του συμφέρον και να δεκτούν να γίνουν ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπενγκαρσία Μπλάνκο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε είπατε εκπρόσωπε, όπως είπατε η Βενεζουέλα και η περιοχή υποφέρουν μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις ε, των καιρών μας. Προβλέπετε μάλιστα ότι θα επιδεινωθεί η κατάσταση με το πέρασμα του χρόνου αν τελικά δεν βρεθεί μια πολιτική λύση. Νομίζω ότι έχουμε δύο αναλύσεις εδώ. Καταρχήν, η διεθνή κοινότητα θα πρέπει να εμπλακεί πολύ περισσότερο, χρειάζονται πολύ περισσότεροι πόροι. Μιλάμε μάλιστα για μια κρίση η οποία μπορεί να συγκριθεί με την ε, συριακή κρίση. Όμως, όπως υπόθηκε και εδώ και νομίζω ότι και από όλους τους ομιλητές, θα πρέπει πολιτικά να επιληθεί η κατάσταση αν θέλουμε να σταματήσει η ανθρωπιστική αυτή καταστροφή και νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά να βρούμε μια ειρηνική λύση για ελεύθερες εκλογές, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν δύο μέρη τελικά και αναγνωρίζοντας και το άλλο μέρος εδώ πρόκειται για την αναζήτηση εναλλακτικών σεναρίων και ε, αυτό δεν λύνεται με το να αυτομαστιγωνόμαστε... αλλά με το να έχουμε θάρρος. Ζητήθηκε εδώ θάρρος και εγώ ζητώ από εσά να είστε θαραλέος κύριε Πατεκπρόσωπε, για να μπορέσουμε να φύγουμε από αυτό το νεκρό σημείο στο οποίο βρίσκεται η Μεζουέλα και να βοηθήσουμε τους πολίτες. Ευχαριστώ η κυρία Κινίτσι για ένα λεπτό. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε είπατε εκπρόσωπε, πριν από πέντε μήνε, εδώ σε αυτή την ίδια αίθουσα, είχαμε μια συζήτηση για την δραματική κατάσταση που πλήττει τη Βενεζουέλα. Και σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε και πάλι στο να συζητάμε το ίδιο θέμα, γνωρίζοντα όμω δυστυχώ ότι με την πάρδο του χρόνου η ε, ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα επιδεινώνεται. Ο αριθμό των προσφύγων και παιδιά ε, ε, αυξάνεται, αυξάνεται συνεχώ. Και για όσου μένουν στη Βενεζουέλα, οι συνθήκε διαβίωση είναι όλο και πιο δύσκολε δεν έχουν τα βασικά, ε, υπάρχουν φαινόμενα βίας. Έτσι λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι όλο και πιο αφόρητο για τον ε, λαϊκό, για τον λαό της Βενεζουέλας να ζει στη χώρα. Πρέπει εμείς ε, να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας, να αναπτύξουμε διπλωματικές προσπάθειες για να στηρίξουμε μια ειρηνική λύση της κρίσης που θα οδηγήσει σε ελεύθερες εκλογές. Βέβαια, εντωμεταξύ πρέπει να προσφέρουμε την απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια για να μην είναι τόσο δυσάρεστη δυσάρεστη η κατάσταση ενός λαού που υποφέρει εδώ και τόσο πολύ καιρό. Ευχαριστώ πολύ κύριο Φιντάνσα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα είναι ε, δραματική. Έχουμε πάρα πολλούς πρόσφυγες ε, οι οποίοι ε, δεν έχουν τίποτα και δεν μιλάει κανείς για αυτούς. Στην Ιταλία έχουμε μια δική μας πρωτοβουλία και αναγνωρίσαμε το δικαίωμα σε Βενεζουελάνους που είναι Ιταλικής προέλευσης να έρθουν πίσω στην Ιταλία. Πρέπει να υπάρξουν ελεύθερες εκλογές. Η Ευρώπη και τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν περισσότερα να σκεφτούν το πώς ε, μπορούν ε, να εντάξουν στις ε, δικές τους τις κοινωνίες όσους θέλουν να επιστρέψουν και είναι προέλευσης ευρωπαϊκής. Δυστυχώς ε, έχουμε πάρα πολλούς ε, πρόσφυγες ε, που έρχονται από την Αφρική, είναι μουσουλμάνοι και υποτίθεται για αυτούς ενδιαφερόμαστε, ενώ για τους άλλους που είναι χριστιανοί και θέλουν να φύγουν από την πατρίδα τους, από ένα κομμουνιστικό καθεστώς, δυστυχώς για αυτούς δεν ενδιαφερόμαστε τόσο πολύ και αυτοί εξαναγκάζονται να ζουν στην πείνα και τη φτώχεια. Ευχαριστώ πολύ τέσσερις ε, βουλευτές που έχουν ζητήσει το λόγο. Χουάν Λόπες Αγγιλάρ πρώτα, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, είπατε εκπρόσωπε Μπορέλ, καλώς ήρθατε. Για μια ακόμη φορά η Βενεζουέλα δεν ε, θα έρθετε εδώ σε κάποια ολομέλεια που να μην υπάρχει μια συζήτηση για τη Βενεζουέλα και πάρα πολλά ε, δεδομένα ανατριχιαστικά ακούμε και ένα μεγάλο μέρος της οικογένειάς μου ζει στη Βενεζουέλα. Είχαμε μετά τον εμφύλιο ανθρώπους που έφυγαν για να βρουν καταφύγιο στη Βενεζουέλα. Όμως ακριβώς μιλάμε για καταφύγιο και θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι από αυτές τα 4,5 εκατομμύρια που έφυγαν από τη Βενεζουέλα ψάχνοντας ε, που να καταφύγουν οι περισσότεροι χτύπησαν την πόρτα της Ισπανίας. Είναι γλαφυρά τα νούμερα. Μεταξύ του 2014 και του 2019 είχαμε ε, ε, αύξηση 100% των αιτήσεων ασύλου στην Ισπανία την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου 4.170 ε, και αφού μιλάμε για αλληλεγγύη θα πρέπει να μιλήσουμε και για αλληλεγγύη σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αιτούντων ασύλου μεταξύ των, μελών, ε, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινώντας από τους Βενεζολάνους που τόσο μας ανησυχούν και τόσο τους αγαπάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Η ε, κυρία για ένα λεπτό. Η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα είναι υπαρκτή και επιδεινώνεται. Ε, βέβαια δεν είναι τυχαία και ούτε είναι απλώ ε, λυπηρή. Δημιουργήθηκε από δεκαετίες προσπαθειών των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσουν ένα σφιχτικό κλειό γύρω από αυτή την χώρα, να καταστήσουν αδύνατο για τον λαό της Βενεζουέλας να αποφασίσει το δικό του μέλλον, να τους εξαναγκάσει στην φτώχεια και στην πείνα. Αυτό οδήγησε στη σημερινή, ανθρωπιστική ε, κρίση. Και φυσικά ο μη εκλεγής ε, Γκουαϊδό ε, φέρνει μόνο ντροπή στο Ευρωπαϊκό Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν προσπάθειες διασπάθησης των κονδυλίων που εσείς λέτε ότι απευθύνονται προς ανθρωπιστική βοήθεια. Μπορούμε να λέμε ότι υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά οι είναι αυτέ ε, που στερούν από του ε, πολίτε ένα ε, δίκαιο μέλλον. Υπάρχουν περισσότερα στοιχεία ανά τον κόσμο που ανήκουν στους Βενεζολάνους. Βοηθήστε τους λοιπόν να ανακτήσουν τα περισσότερα του στοιχεία για να τους βοηθήσουμε να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Μπορέλ, είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε προβλέψει 320 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη της Βενεζουέλας και είμαστε διατεθειμένα να κάνουμε περισσότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Αμερικανικό τραπεζικό κλάδο έχουν εκλέψει δεκάδε δισεκατομμύρια δολάρια από του Βενεζολάνου. Αν θέλετε λοιπόν να κάνετε περισσότερα, πρέπει να του βοηθήσετε να ανακτήσουν τα χρήματά του. Να αρθούν οι κυρώσει. Μα γιατί στο καλό η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίζει αυτές τις παράνομες αμερικανικές κυρώσεις. Δεν υπάρχει καμία λογική. Καταστρέφουν τη χώρα. Ε, ο Μαδούρο δεν είναι κανένα καταπληκτικό ε, ηγέτη ενδεχομένω, αλλά δεν ξέρω και πολλού τέτοιου ε, χαρισματικού όλο τον κόσμο. Η σημερινή κρίση έχει προκληθεί από τι μερκανικέ κυρώσει μία από τις ε, πιο φημισμένες ε, ευρωπαϊκές ε, νομικές εταιρείες στο Παρίσι αμφισβητεί ακριβώς τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Βενεζουέλα και προσπαθεί να ανακτήσει κάποια από αυτά τα χαμένα προσωπικά στοιχεία. Σας παρακαλώ λοιπόν να διαδραματίσετε σημαντικό και ενεργό ρόλο για την άρση αυτών των κυρώσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φάβιο Καστάλντο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρά την προσοχή των, ε, το ότι η προσοχή των ΜΜΕ έχει στραφεί σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί στη στη Βενεζουέλα και σήμερα αποτελεί την πιο ανησυχητική κρίση οι Βενεζουλάνοι συνεχίζουν ε, να υφίσταται όλο και πιο σοβαρές ε, συνέπειες μια πρωτοφανούς οικονομικής ε, κρίσης στη Λατινική Αμερική. Πρόκειται για μια χρόνια κρίση και είναι δύσκολο να δούμε το τέλος της και έχουμε και μια πολιτική κρίση που έχει προσθεθεί. Πρέπει όμως να ξεπεράσουμε τον οπορτουνισμό και να εργαστούμε από κοινού προκειμένου να προσφέρουμε ανακούφιση στον πληθυσμό της Βενεζουέλας που ζει καθημερινά σε μια επίγουσα κρίση ανθρωπιστική. Θα πρέπει να συντονιστούμε για να υποστηρίξουμε τις 16 χώρες ε, που ε, τις αφορά η κρίση και έχουν ε, υποδεχθεί τους μετανάστες από τη Βενεζουέλα. Η διάσκεψη που έγινε στις Βρυξέλλες είναι σημαντικό βήμα ε, για να ακολουθήσουμε και να δώσουμε συνέχεια στη διαδικασία του Κίτο. Και ε, εν ώψη και μιας δεύτερης διάσκεψης ας, ακούσουμε, ας κάνουμε συγγνώμη τη φωνή μας να ακουστεί. Thank you. I give the floor. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό τους εκπρόσωπους της Ένωσης, για τα καταληκτικά, καταληκτικά του σχόλια. Κύριε Μπορέλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλοι υπενθυμίσατε και περιγράψατε μια κατάσταση που είναι γνωστή. Είναι προφανές ότι έχουμε ένα πολιτικό πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να με πείσετε γι' αυτό. αλλά εγώ προσωπικά έχω ένα θέμα συνείδησης. Φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς ε, μπορεί να έχετε το ίδιο. Γιατί είναι προφανές ότι παρόλα όσα αυτά μπορούμε να πούμε για το καθεστώς Μαδούρο, αυτή η χώρα δεν έχει την δυνατότητα να αξιοποιήσει τους οικονομικούς της πόρους. Από το 2017, εξαιτίας ε, των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί, η Βενεζουέλα ε, δεν κατάφερε να εξαγάγει 400.000 ε, βαρέλια την ημέρα από το πετρελαιό της. Αυτό μεταφράζεται σε 8 δις δολάρια τέσσερις φορές το ποσό των ε, εισαγωγών τροφίμων. Και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και αν συνεχίσουν να πέφτουν ε, τα έσοδα από το πετρέλαιο κατά 60% όπως προβλέπετε, θα έχουμε επιπλέον 300.000 άτομα που δεν θα έχουν πρόσβαση ούτε στην τροφή ούτε στα φάρμακα. Πρέπει να είναι κανείς τυφλός για να μην ε, κατανοήσει ότι τα εκατομμύρια των ε, προσφύγων οφείλονται σε αυτό το γεγονός, ότι η χώρα δεν μπορεί να αξιοποιήσει τους σπόρους της. Αυτό βέβαια δεν εξηγεί την ε, πολιτική κριτική κατά του καθεστώς Μαδούρο. Ο κύριος, κύριε Ταγιάννη, όχι, καθόλου δεν ε, αποτελεί δικαιολογία αυτό. Δεν αποτελεί δικαιολογία. Δεν είναι προφανές όσο κομμουνιστής και αν είναι ο δικτάτορας ε, ότι ο αντίκτυπος ε, κάποιων κυρώσεων δεν μπορούμε να τον αρνηθούμε τον αντίκτυπο και στην πολιτική κρίση προστίθεται και μια ανθρωπιστική κρίση και δεν μπορούμε να περιμένουμε να δώσουμε λύσεις σε αυτό <laughs> μέσω της διεθνούς κοινότητας η οποία φιλανθρωπικά θα δίνει πόρους γιατί δεν είναι δυνατόν να θρέψουμε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους καθημερινά δεν είναι δυνατόν ε, να βρούμε τόσους πολλούς ανθρωπιστικούς πόρους. Το πολιτικό πρόβλημα είναι ένα και δεν ε, χρειάζεται κανένας να με πείσει ότι είναι απαραίτητο να γίνουν ε, τα πάντα για να υπάρξουν εκλογές στην ε, Βενεζουέλα. Δεν χρειάζομαι διδάγματα, όμως ούτε μπορούμε να αρνηθούμε μια πραγματικότητα και πολλοί από εσά το είπατε. Πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις που να επιτρέψουν σε μια γιγάντια ανθρωπιστική κρίση ε, που είναι συνέπεια του καθεστώτος να επιληθεί. Εσείς ψηφίσατε εδώ διάφορα ψηφίσματα όπου είπατε ότι καμία κύρωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί εάν ε, πλήττει το λαό της Βενεζουέλας. Αυτά τα ψηφίσατε εσείς. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εφαρμόσει οικονομικές κυρώσεις ε, κατά του λαού της Βενεζουέλας, αλλά κατά των ηγετών, κατά των κυβερνώντων και αν χρειαστεί θα επιβάλλουμε και άλλες αλλά κατά των κυβερνώντων. Δεν μπορείτε να αναμένετε να επιληθεί η κρίση της Βενεζουέλας καταδικάζοντας ε, μαζικά στην πείνα τον πληθυσμό. Είναι ένα σοβαρό πολιτικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με πολιτικό τρόπο. Δεν μπορούμε όμως να κλείνουμε τα μάτια στην αναγκαιότητα και πολλοί το είπαν να αναζητήσουμε λύσεις που να αντικαθιστούν ε, μια ανθρωπιστική ε, βοήθεια που δεν θα δώσει η διεθνής κοινότητα γιατί δεν ε, μπορούμε να συγκεντρώσουμε τόσα δισεκατομμύρια που χρειάζονται σε δωρεές. Τώρα μιλάμε ουσιαστικά για κάποιες εισφορές που δίνονται που είναι 10 φορές αυτή η ποσότητα. Έχουμε λοιπόν ένα τεράστιο πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο δικτάτορας είναι ο κομμουνιστής. Το πρόβλημα είναι ότι η χώρα αυτή βρίσκεται σε μια δύσκολη πολιτική κατάσταση, στην οποία πρέπει να απαντήσουμε και όπως πράττουμε και νομίζω ότι έχει ενεργοποιηθεί πολιτικά και διπλωματικά η Ευρώπη γι' αυτό, αλλά δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια ότι λαμβάνονται μέτρα αντίθετα από αυτά που ψηφίσατε εσείς. Έχουν ληφθεί μέτρα που ζημιώνουν ε, δραματικά το λαό της Βενεζουέλας. Και πιστέψτε με, αυτή δεν πρόκειται να είναι η λύση. Δεν μπορεί να αποτελέσει αυτό τη λύση. Παρακαλώ αφήστε τον ομιλητή να εκφραστεί. Νομίζω ότι πρέπει να σεβαστείτε τους κανόνες. Εδώ. Θα προσπαθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει τους διπλωματικούς ε, και πολιτικούς της ε, διάβλους σε πλήρη συνεργασία με την κυρία Μπασελέ. Φυσικά ε, δεν αέρουμε τις ευθύνες ε, από το καθεστώς της Βενεζουέλας, όμως ε, θα ήταν λάθος να σκεφτούμε ότι θα μειωθούν οι μεταναστευτικές ροές. Αν, ε, συνεχίζεται να, αν συνεχιστεί η οικονομική ασφυξία στη χώρα. Thank Ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει στην επόμενη ολομέλεια επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι δήλωση του είπα εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την ανθρωπιστική κατάσταση και τη δημοκρατία στην Ικαράγουα και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μπλε κάρτες ε, με ηλεκτρονικό σύστημα. Ε, οι σχετικές οδηγίες υπάρχουν ε, μπαίνοντα στην αίθουσα της Ολομέλειας. Και επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι οι ερωτήσεις μπλε κάρτας μπορούν να γίνουν μόνο μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών των Ευρωβουλευτών. Και η ε, συζήτηση ξεκινάει με τον κύριο Μπορέλ. Παρακαλώ κύριε Μπορέλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, εξότιμα μέλη, η κατάσταση στην Ικαράγουα ε, συνεχίζει να εμπνέει μεγάλη ανησυχία. Είναι μη βιώσιμη. Η στάση Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι συνεπής από την αρχή της κρίσης. Η πολιτική μας είναι να στηρίξουμε μία ειρηνική διαπραγμάτευση και δημοκρατική λύση πάνω απ' όλα. Όπω και στην περίπτωση τη Βενεζουέλα, μόνο ο λαό τη Νικαράγουα μπορεί να διαλέξει του ηγέτε τη και του εκπροσώπου τη σε ελεύθερε και δίκαιε εκλογέ. Ακριβώ τα ίδια ισχύουν και με τη Βενεζουέλα, λοιπόν, εδώ. Η κυβέρνηση πρέπει να σέβεται και να υπερασπίζεται τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών τον περασμένο Ιανουάριο, ακριβώς πριν από την ε, επίσκεψη του Κοινοβουλίου στη Μανάγουα, το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων υπογράμμισε τη βούλησή του να αξιοποιήσει όλα τα μέσα πολιτικής ε, προκειμένου να υπάρξει μια ειρηνική λύση στην κρίση και για να μην υπάρξει περαιτέρω υπονόμευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στις αρχές ε, του έτους, η κυβέρνηση της Νικαράγουα ε, δέχθηκε να βρεθεί μία λύση και υπέγραψε ένα προσωφωνητικό για την απελευθέρωση ε, πολιτικών κρατουμένων και για την ε, επαναγκατάσταση κάποιων θεμελιωδών ελευθεριών. Όμως βλέπουμε ότι αυτό δεν συνέβη τελικά. Πολλοί απελευθερώθηκαν και αμέσως μετά συνελήθησαν εκ νέου. Και δεν έχουν υπάρξει εκ νέου οι πολιτικέ ελευθερίε που απαιτούνται. Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων υιοθέτησε ένα πλαίσιο για μεμονωμένε και στοχευμένε κυρώσει στα μέσα Οκτωβρίου. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά. Απαγορεύεται η είσοδο στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια και παγώνουμε τα περιουσιακά στοιχεία ατόμων ή οργανώσεων που έχουν διδραματίσει ρόλο κλειδί στις παραβιάσεις ανθρωπινών δικαιωμάτων από το καθεστώς. Οι κυρώσεις λοιπόν είναι μεμονωμένες, αναστρέψιμες και πάνω απ' όλα ε, στοχεύουν, στην, ε, μάλλον, στοχεύουν στο να μην πλήξουν ε, τον λαό της Νεκαράκος, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο. Σε τρει τομείς πρέπει να υπάρξει απτή πρόοδος, προκειμένου να διαμορφώσουμε τις προποθέσει για μια ειρηνική και δημοκρατική έξοδο από την κρίση έχουν να κάνουν με τις ε, δεσμεύσει που έχει αναλάβει η ίδια κυβέρνηση. Δεν απαιτούμε κάτι παραπάνω. Θέλουμε απλώς να τηρήσει τις δεσμεύσει τη. Συστηματικά έχουμε επαναλάβει και δημόσια και κατηδίαν κάτι το οποίο έχει συμπεριληφθεί και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου τον περασμένο Οκτώβριο και συνάδει ε, με τις συστάσεις ε, που έχουν εκδοθεί πρόσφατα Πρώτον, θέλουμε την θέσπιση πολιτικών ελευθεριών και το νομικό καθεστώς ε, των απαγορευμένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και απελευθέρωση των ε, πολιτικών κρατουμένων και πλήρη απαλλαγή τους από τις κατηγορίες. Δεύτερον, πλήρη συνεργασία και επιστροφή των ε, φορέων, των διεθνών φορέων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μεταξύ αυτών και το γραφείο του ΙΣΥΠΑ της Αρμοστία για Θεμελιώδη Δικαιώματα και την ε, Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπινών Δικαιωμάτων. Τρίτον, συμφωνία για την εκλογική μεταρρύθμιση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Μαζί και με την Syndical ε, Alliance. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, λοιπόν, θα πρέπει να διαμορφωθεί το εκλογικό σύστημα και να συνάδει και με τις συστάσεις των εκλογικών παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε διατεθειμένοι να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια με την εμπειρογνωμοσύνη της, ενδεχομένως και με αποστολή εκλογικών παρατηρητών. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο πλευρό του λαού της Νικαράγουας και επιθυμίζει ότι πρέπει να σταματήσει η καταστολή και θα πρέπει να επανέλθει και να διασφαλιστεί ο σεβασμός ε, προς τα συνταγματικά δικαιώματα όλων των πολιτών. Μεταξύ αυτών η ελεύθερη η ελευθερία έκφρασης, ε, το δικαίωμα του συνέρχεστε, συναθρίζεστε ε, και οι ειρηνικές διαδηλώσεις. Αυτά ήθελα να τονίσω εκ νέου ενώπιόν σας και ελπίζω με την στήριξή σας να ασχίσουμε περισσότερη πίεση για να πετύχουμε αυτές ακριβώς τις δεσμεύσεις μας. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Λόπες Χίλ, εκ μέρους του ΕΛΚ, για δύο λεπτά. Θα ήθελα να χαιρετήσω τα λόγια του είπα του εκπροσώπου η κρίση στην Νικαραγώγα ξεκίνησε από την ε, υψηλή συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια των Ορτέγα. Η καταστολή της αντιπολίτευσης της κοινωνίας των πολιτών, των δημοσιογράφων και της κοινωνίας ε, γενικά ε, έλαβε χώρα. Ο στραγγαλισμός του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας συνοδεύεται από ατιμορρησία και από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θυμηθούμε σήμερα ότι δεν ε, υφίσταται ε, μόνο οι κάτοικοι της Νικαράγουας ε, κάποιες κυρώσεις, αλλά και Ευρωπαίοι. Έχουμε την Αμάγια Κόπενς, η οποία συνελήφθη το 2018 επειδή συμμετείχε σε ειρηνικές διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος και βρίσκεται ξανά σήμερα στη φυλακή επειδή βοήθησε κάποιες γυναίκες που ήταν σε απεργία πείνας. Όταν εκτάσαμε την ε, δέκατη επέτειο τη ε, Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, και είπαμε ότι η Ευρώπη είναι το λίκνο αυτών, ε, θα πρέπει να έχουμε κατά νου τους ανθρώπου που υπερασπίζουν τι αξίε μα και γι' αυτό βρίσκονται στη φυλακή. Το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να ξεχάσει του Ευρωπαίου πολίτε που υποφέρουν στα χέρια σκληρών δικτατοριών επειδή υπερασπίζουν τι αξίε μα, την ελευθερία, τη δημοκρατία, καταπολεμούν την ανισότητα και υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Μάγια Κόπενς δεν είναι η μόνη, δυστυχώς, ε, και γι' αυτό θα πρέπει να υψώσουμε τη φωνή της Ευρώπης μέχρι να απελευθερωθούν όλοι αυτοί. Σας ευχαριστώ. κυρία Λετάο Μάρκε από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πετεκπρόσωπε. Για μια ακόμη φορά αυτό το κοινοβούλιο έχει εκδηλώσει την ανησυχία του με την πολιτική κατάσταση στην Ικαράγουα τονίζοντας τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις ε, ε, συλλήψεις ε, χωρίς λόγο και την ανυπαρξία στο δικαίωμα της ενημέρωσης. Πρόσφατα κάποιοι ακτιβίστες ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, όπως και η Αμάγια Εύα Κόπενς ε, συνελήφθησαν επειδή μοίραζαν νερό και φάρμακα σε μητέρες συλληφθέντων που βρίσκονταν σε απεργία πείνας στην εκκλησία του Αγίου ε, Μιχαήλ στη Μασάγια. Ε, μάλιστα μάθαμε ότι η κυβέρνηση Νικαράγου έχει εντατικοποιήσει τη δίωξη κατά όλων ε, των ακτιβιστών και των οικογενειών τους που τοποθετήθηκαν κατά των πολιτικών της και γι' αυτό εκ νέου εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας με τον λαό της Νικαράγουας και ζητούμε από το Συμβούλιο να ε, υιοθετήσει κυρώσεις ε, παγώματος των περιουσιακών στοιχείων και της απαγόρευσης χωρίς θεωρήσεων σε όσους είναι υπεύθυνοι για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενθαρρύνουμε την κυβέρνηση Νικαράγουα να ξανά ε, αρχίσει το διάλογο με την Αλιάνσα Σίβικα για να βρεθεί μια λύση σε αυτή τη σύγκρουση, να διαλύσει τις παραστρατιωτικές οργανώσεις, να υποστηρίξει τη μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος, να απελευθερώσει τους πολίτες που κρατούνται παράνομα και να ξαναδώσει ε, νομικό και προσωπικότητα στις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Επίσης, ε, ζητάμε από τον ύπατο εκπρόσωπο και από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυ στην κατάσταση αυτή και ζητάμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στείλει μια αντιπροσωπεία στην Ικαράγουα το συντομότερο. Όλοι μας ε, που αντιστεκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση στην Ικαράγουα ε, όλοι μάλλον όσοι αντιστέκονται στην Ικαράγουα πρέπει να ξέρουν ότι δεν θα αγνοήσουμε τον αγώνα τους ούτε θα τους εγκαταλείψουμε στη μοίρα τους. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Νάρτ για δύο λεπτά το Ρινιού είμαι κύριε Μπορέλ, υποστηρίζω την ομιλία σας ε, ως ρεαλιστική και απαραίτητη. Θέλω να υπενθυμίσω ότι το 1979 ο λαός της Νικαράγουας αγωνίστηκε για την αξιοπρέπεια, την ελευθερία και τη δημοκρατία κατά της δικτατορίας του Σομόσα. Εγώ ήμουν εκεί και θυμάμαι ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Φελίπε Κονσάλες είχε υποστηρίξει ε, τον ε, αγώνα αυτών. Και τόσα χρόνια μετά βλέπουμε ότι ε, υπάρχει ουσιαστικά καταπίεση των δικαιωμάτων από ε, το ζευγάρι Ορτέγα Μουρίγιο. Σήμερα έχουμε τις ένοπλες ε, συμμορίες και την αστυνομία που δολοφονούν τους ανθρώπους. Η Διεθνής Αμνηστία και η Human Rights Watch, ο ΙΕ, είναι ε, κατηγορηματικές ε, γιατί στην Ικαράγουα δεν υπάρχει ούτε δικαιοσύνη, ούτε δημοκρατία, ούτε ανθρώπινα δικαιώματα. Βασικές ε, αρχές που δεν μπορούν να αποκλείονται από την συνείδησή μας και την αλληλεγγύη μας. Γι' αυτό οι πιο μεγάλες ομάδες στο Κοινοβούλιο συμφώνησαν σε ένα κοινό ψήφισμα χωρίς τροπολογίες αποκλείστηκαν, αυτοαποκλείστηκαν μάλλον μόνο ε, όσοι έχουν ε, ιδεολογικά σύνορα. Εμείς θέλουμε να δηλώσουμε την ελεγγύη μας με τους βασανισμένους και με τους εξαφανισμένους και με όλο το λαό της Νικαραγωγής. Περάσουμε στις πράξεις. Η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεντρικής Αμερικής βασίζεται ε, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γι' αυτό θα έχουμε στο ψήφισμα σημαντικά στοιχεία το να προωθήσουμε μια δημοκρατική λύση μέσω αξιόπιστων εκλογών που θα οδηγήσουν σε σημαντική μεταρρύθμιση του συστήματος ε, και της ε, ε, δικαιοσύνης Η αποστολή αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ικαραγωγούμενη στην πρώτη με τον Ραμόν Χαουρέγγι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτήσει έναν κατάλογο ανθρώπων στους οποίους θα επιβληθούν κυρώσεις και να ενεργοποιηθεί το άρθρο αναστολής που υπάρχει στη Συμφωνία Σύνδεσης. Η κυρία Μέντς, εξ των Πρασίνων, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, τους τελευταίους μήνες ε, ο πληθυσμός της Νακαράγκος αντιμετωπίζει κυβερνητική καταστολή. Είχαμε πολυάριθμες παρεμβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Εκατοντάδες έχουν συλληφθεί παράνομα για ειρηνικές ε, διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης, μεταξύ αυτών και η Βελγίδα Αμάγια Κόπενς. Πρόκειται λοιπόν για παραβιάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις ε, αρχές και καλούμε τις αρχές της Νικαράγουα να σταματήσει ευθύ αμέσω ε, την καταστολή κατά του λαού τη. Θα πρέπει να υπάρξουν ελεύθερε και δημοκρατικέ εκλογέ το σύντομα δυνατόν. Οι διπλωμάτε μα στην Νικαράγουα θα πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλουν προσπάθειε για να συμφιλειώσουν ε, τι διαφορετικέ πλευρέ και να στηρίξουν ε, τα κινήματα της κοινωνίας των πολιτών, χωρίς όμως να λαμβάνουν μια κυρίαρχη δεσπόζουσα θέση. Η λύση δική μας είναι ένα συμβασμός μεταξύ διαφορετικών κομμάτων. Υπάρχουν ζητήματα που είναι σημαντικά για μας τους πράσινους ε, και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο κοινό κείμενο. Για παράδειγμα, η ευθύνη των ευρωπαϊκών εταιριών και ο ρόλος τους στην σταθεροποίηση αυτής της ε, ακανθόδους ε, κυβέρνησης. Πρέπει λοιπόν να δούμε και τις, ε, τα πεπραγμένα των ευρωπαϊκών εταιριών στην Νικαράγουα και τα μέτρα δέσους επιμέλειας που λαμβάνουν. Σε περίπτωση ε, συνενοχής, σε περίπτωση παραβίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα πρέπει και αυτές να λογοδοτήσουν. Ως Πρόεδρος της ε, Αντιπροσωπείας για την Αμερική ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτό το ψήφισμα γιατί πρόκειται για ένα σημαντικό μήνυμα αλληλεγγύη προς το λαό της Νικαράγουα, που αντιμετωπίζει παραβιάσεις των θεμελιωδών του δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Mr. Terch. Ο κύριος Τέρτ, εκ του ΙΣΙΑΡ, e για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Μπορέλα, η κτηνοδία του σοσιαλιστικού καθεστώτος την ελορτέγα στην Ικαράγουα συνεχίζει ε, να ε, προκαλεί τρόμο και νεκρούς και μέχρι τώρα ήταν άχρηστες ε, όλες οι προειδοποίησεις που έγιναν από το εξωτερικό για να σταματήσει το καθεστώς αυτό το σπιράλ μαζικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, δηλαδή τίποτα δεν χρησιμεύσε και τώρα είχαμε στη τελευταία κρίση εκατοντάδες δολοφονίες μαζικά βασανιστήρια εξοδικαστικές εκτελέσεις το ίδιο σενάριο που είδαμε και στην Βενεζουέλα γιατί στην πραγματικότητα μιλάμε για δύο παράλληλα, δύο ίδια καθεστώτα, τα οποία διέπονται από την ε, ίδια σκληρή αυθαιρεσία, η ε, ε, οποία προέρχεται και δίνεται κατεύθυνση από την Κούβα. Δηλαδή, συνεχίζουμε να γνωρούμε ότι η Κούβα προστατεύει την Νικαράγουα και τη Βενεζουέλα και προστατεύει αυτή την εγκληματικότητα που βλέπουμε τώρα στη Λατινική Αμερική. Ελπίζω να αντιδράσετε. Ο κύριος Ορμπάν Κρέσπο, εκ μέρους της Γκουέντζιελ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το να καταγγέλουμε την ε, καταστολή κατά του λαϊκού κινήματος από την Σορτέγα Μωρίγιο ε, δεν σημαίνει ότι πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι των οικονομικών ελίτ της Νικαράγουα στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να υποστηρίξει μια πολιτική λύση που να περνά από την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, την πάυση της βίας και την αναγνώριση του ρόλου των κοινωνικών κινημάτων στις διαπραγματεύσεις. Μην κάνουμε λάθος. Ε, όταν ε, πολλοί από τους βουλευτές ασκούν κριτική στον Ορτέγα δεν το κάνουν επειδή ανησυχούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά για τα οικονομικά συμφέροντα των Ευρωπαίων πολυεθνικών των Ευρωπαϊκών Πολυεθνικών, όταν εμεί ασκούμε κριτική στην κατάσταση στην Καράκουα, υπερασπίζουμε, ε, πρέπει να υπερασπίσουμε το λαό στο να οικοδομηθεί ε, μια αλλαγή προκειμένου να ακολουθεί το πνεύμα τη Ανδυνιστική Επανάσταση που τόσε ελπίδε δημιούργησε στι λαϊκέ τάξει σε ολόκληρο τον κόσμο. Mr. Ο κύριος Σόιδο ε, Άλβαρες, για ένα μισή λεπτό. Πρόεδρε, κύριε είπατε εκπρόσωπε, αύριο θα εγκρίνουμε ένα ψήφισμα, θα ψηφίσουμε μάλλον ένα ψήφισμα όπου καταγγέλουμε εκ νέου τις σοβαρές παραβιάσεις που λαμβάνουν ε, χώρα σε ό,τι αφορά το σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στην Ικαράγουα. Δυστυχώς η κατάσταση δεν βελτιώθηκε, το αντίθετο Μάλιστα, ε, τίθεται σε κίνδυνο και το κράτος δικαίου και τα νούμερα είναι ενισχυτικά. Πάνω από 80.000 ε, άτομα εγκατέλειψαν ε, την Νικαράγουα και περίπου άλλοι 300 έχουν δολοφονηθεί. Εκατοντάδες βρίσκονται υποκράτηση. Εκατοντάδες φοιτητέ, εκδιώθηκαν από το Πανεπιστήμιο και εκατοντάδες δημοσιογράφοι έπρεπε να εγκαταλείψουν τη χώρα λόγω της καταστολής που ασκεί η κυβέρνηση της Νικαράγουα η δημοκρατική αντιπολίτευση και η κοινωνία των πολιτών βρίσκονται σε μια φόρητη κατάσταση. Τι άλλο θα πρέπει να γίνει για να επιβάλλουμε κυρώσει σε αυτού που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε μια χώρα τέρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ έχουμε συμφωνία σύνδεση μαζί του. Κύριε Πατακπρόσωπη, γνωρίζετε καλά ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο λαό στην Καράγουα είναι αξιοθρύνητη. Και καθώς ε, επιδεινώνεται συνεχώς ε, η κατάσταση, ε, τι θα πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν μπορούμε να απογοητεύσουμε το λαό της Νικαραγώ, γι' αυτό ζητάμε άμεση απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, το να σταματήσει η καταστολή της αντιπολίτευσης, να μπορέσουν να ασκηθούν οι θεμελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Λόπες, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον είπα το εκπρόσωπο, τον κύριο Μιζομπορέλ. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να καταγγείλουμε την σοβαρότατη κατάσταση στην Ικαράγουα σε ό,τι αφορά την παραβίαση των δημοκρατικών δικαιωμάτων που είδαμε τους τελευταίους μήνες και χρόνια στη χώρα και μάλιστα βλέπουμε όλο ένα και μεγαλύτερη εχθρότητα της κυβέρνησης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε ότι ότι συλλήψεις ε, φοιτητών, ε, κοινωνικών ηγετών και ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων λάμβαναν χώρα στην Καράγουα. Και πρέπει να αναφέρουμε και την περίπτωση της Αμάγια Κόπενς. Ε, μάλιστα, ακούσαμε και βασανιστήρια κατά τη διάρκεια των συλλήψεων αυτών. Ε, και θα πρέπει να ζητήσουμε την άμεση απελευθέρωση όλων αυτών των κρατουμένων. Ζητάμε και ένα κατάλογο κυρώσεων για να κάποιους ε, ε, ανθρώπους που συμμετέχουν στην κυβέρνηση για να βρούμε μια διέξοδο, μια ειρηνική δημοκρατική διέξοδο που θα εγγυάται το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και που θα διασφαλίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμμετέχει στη δημοκρατική μετάβαση στην Καράγου. Η κυρία Μπιλμπαουεραντίκα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η Νικαράγουα ε, θα πρέπει μάλλον ξεκίνησε την κρίση της από το Μάρτιο του 2019 θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η σανδινιστική κυβέρνηση, σύμφωνα με τελευταία στατικά στοιχεία, έχει προκαλέσει 328 θανάτους. Αν συνεχιστεί ε, το λοκάρισμα, εγώ υποστηρίζω τις ε, κυρώσεις κατά αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων κατά του Ορτέγα και της ε, Μουρίγιο. Χρειάζεται να ασκηθεί πολιτική στην κρίση αυτή. Γι' αυτό ζητούμε από τον Ορτέγα να συγκρίνει την πρώτη του φωτογραφία της 1η Ιανουαρίου του 1985 όταν ορκίστηκε με αυτές που βγάζει σήμερα. Σήμερα έχουμε μια αξιολύπητη κατάσταση και ε, τίποτα δεν μοιάζει με την ελπίδα που είχαμε όταν βγήκε η χώρα από τη δικτατορία του όμως 80.000 άνθρωποι έφυγαν από την Βεζουέλα και αρχίζουν ε, να σκέφτονται ε, ότι έχουν δύο, υπάρχουν δύο πολύ διαφορετικές πορείες που αρχίζουν όμως να μοιάζουν πάρα πολύ. Η κυρία Κάνκο για ένα λεπτό. <laughs> Uh, Ο Μάρτε Μέσμακερ, που είναι στο κόμμα μου, ε, στην αρχή της χρονιάς έψαξε και αναζήτησε την Αμάλια Κόπενς Υπάρχουν ε, χιλιάδες φοιτητές ε, στη φυλακή στη Μαναγουά γιατί διαδήλωσαν κατά της κυβέρνησης Ορτέγα. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν φυλακιστεί στην Εγκαράγουα επειδή βγήκαν στους δρόμους για μια ελεύθερη και δημοκρατική πατρίδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι δημοκρατικέ ελευθερίε. Ε, συχνά ξεχνάει ο κύριος Ορτέγα ότι και αυτός βρέθηκε στη φυλακή επειδή διαδήλωνε και αρνείται να φέρει εις πέρα στις δεσμεύσεις του, του, της από τις αρχές του χρόνου. Εμείς ζητούμε από την κυβέρνηση Ορτέγα να ξεκινήσει το διάλογο και να θέσει τέλος στην συνεχιζόμενη καταστολή. Θα πρέπει να επανέλθει η δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Εγώ θα εξακολουθήσω να παλεύω για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά είναι τα λόγια της Αμάγια Κόπενς όσοι ε, βρίσκονται στη φυλακή εξαιτία των διαδηλώσεων πρέπει να αποφυλακιστούν ε, απευθεία, όπως και αυτή η 25χρονη κοπέλα. Πρέπει να τους βοηθήσουμε. Mrs. Daly, one minute. κυρία για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κάθε μήνα που ερχόμαστε εδώ καταδικάζουμε κάποια εκλεγμένη κυβέρνηση στη Λατινική Αμερική που προσπαθεί να επιβιώσει παρά τις παρεμβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, να καταδικάζουμε τους δράστες. Εγώ τα βρίσκω όλα αυτά τραγικά γιατί είναι οι άνθρωποι σε αυτές τις χώρες που υποφέρουν. Αυτή είναι μια χώρα ε, όπου το 2018 ε, μπόρεσε να αποτρέψει τη βία, ε, μπόρεσε να επιβιώσει παρά τις μονομερείς, τη μονομερή επιβολή κυρώσεων από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Πρέπει λοιπόν ε, να κάνουμε, να συμφωνήσουμε όλοι ότι όλοι επιθυμούν την αποσταθεροποίηση. Η Νικαράγουα και η Κούμπα θα είναι τα επόμενα θύματα. Ο Μοράλε έχει εκδώσει μία δήλωση σχετικά με το παράνομο Καθεστώ στην ε, Νικαράγουα και τελικά η μικρή Νικαράγουα ε, παρουσιάζεται ω μία μεγάλη απειλή στην ασφάλεια των ΗΠΑ. Είναι μία χώρα υποκατάληψη. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να λέμε τα πράγματα με το όνομά του και να αφήσουμε του κατοίκου τη Νικαράγουα να επιλέξουν μόνο του τη μοίρα του. Η κυρία Αρένα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η Νικαράγουα διέρχεται μία πολιτική κρίση εδώ και 1,5 χρόνο. Οι δηλώσει κατά τη κυβέρνηση Ορτέγα, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018, οδήγησαν σε 300 νεκρούς, 2.000 τραυματίε και χιλιάδες φυλακισμένου, όπως και η Μάγια Κόπεν, που ήθελε απλώς να πάει νερό ε, σε κάποιου απεργού πείνα. Η κυρία Μπασλέ το 2017 στην έκθεσή τη ε, είχε αναδείξει τα πολύ σημαντικά παραπτώματα σε ό,τι αφορά τι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθερία έκφραση, ελευθερία ε, συναθρίζεστε υπάρχουν ανεξάρτητα μέσα ενημέρωση τα οποία έχουν κλείσει, έχουν συλληφθεί οι δημοσιογράφοι ε, και οι ηγέτε των αυτόχθονων λαών επίση έχουν φυλακιστεί και το δικαστικό σώμα στερείται ανεξαρτησίας. Θέλουμε λοιπόν την απελευθέρωση. Οδηγεί, μάλλον αναγκάστηκε το, η κυβέρνηση να απελευθερώσει 400 ε, πολιτικούς αυτομένους, αλλά υπάρχουν και άλλοι που πρέπει να αποφυλακιστούν. Όμω η αποκατάσταση τη εμπιστοσύνη θα πρέπει να περάσει από, την, ε, ε, από τον αγώνα κατά τη ατιμορρησία. Γιατί έχουμε πρακτικέ βασανιστήριων και δολοφονιών και οι υπεύθυνοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Χρειαζόμαστε διεθνείς παρατηρητές ε, και χαιρετίζουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Οκτωβρίου. Χρειαζόμαστε στοχευμένε κυρώσει και το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και θα σα στηρίζει στα διαβήματά σα. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, κύριε Ροδρίγε Ράμο. Ευχαριστώ. Κύριε Πατέ, πρόσωπε ο πρόεδρο Ντανιέλ Τοβέ και η σύζυγό του αντιπρόεδρος κυρία Ρωσαρίου Μουρίγιο οδηγούν σε αδιέξοδο την Ικαράγουα, την νοσιογράφη, αντιπολιτευόμενοι, ακτιβιστές, καταστέλλονται με Βία. Έχω εδώ μία επιστολή συγγενών που λέγονται Αγουαδόρας, οι οποίες απήχθησαν και ε, φυλακίστηκαν επειδή πήγαιναν νερό σε 11 μητέρες που βρίσκονταν στην εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ για να ζητήσουν την απελευθέρωση των παιδιών τους. Σε αυτήν την επιστολή λέει ότι μία, η Ελιζαμπέτ Νέιμα είναι πολύ σοβαρά ε, ασθενής, είναι 25 χρονών και της αρνήθηκαν την περίθελψη. Και η Όλγα Μάγερ Σολάρμα Ουρτάδο, Ιβάν Άλβαρε, η Αμάγια Κόπεν και η Γουέντι Χουάρεν ξεκίνησαν την περασμένη Κυριακή απεργία πείνα για να ζητήσουν για φαρμακευτική περίληψη. Οι γονεί τη Νέιμα δεν ξέρουν που βρίσκεται η κόρη του, τους, όπω και δεν το ξέρουν και πολλοί γονεί στην Νικαράγουα. Αλλά αυτό που ξέρουν είναι ότι οι πολιτικοί κρατούμενοι στην Νικαράγουα βρίσκονται ε, σε απάνθρωπε συνθήκε στι φυλακέ ε, και υφίσταται βία. Γι' αυτό απαιτούμε την άμεση επελευθέρωση των κρατουμένων και επιβολή κυρώσεων κατά των υπευθύνων, ξεκινώντας από τον Ορτέγα. Κύριε Χομσχινέλ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εννιά μήνε μεταξύ από τον ε, τελευταίο ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο για την Καράγουα δεν βελτιώθηκε. Ε, η κατάσταση στη χώρα, η καταστολή αυξήθηκε και περιορίστηκαν οι ελευθερίε ε, των πολιτών. Μπροστά σε αυτήν την επιδείνωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα οι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κατοίκων των πολιτών τη Νικαραγουά πρέπει να σταματήσουν αμέσω. Όλοι συμφωνούμε ότι αυτό το ψήφισμα ε, θα πρέπει να πάει πιο μακριά και να θετήσουμε μια πιο σκληρή στάση. Σε προηγούμενα ψηφίσματα το κάναμε και τώρα πρέπει